Καλή σας μέρα! Ακολουθεί η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα τη διανομή τροφίμων στα πλέον άπορα άτομα της Ένωσης. Το λόγο έχει ο Επίτροπος, κύριο Σολιρέν. Uh, Πρόεδρε. Σημειώνω το πόσο σημαντικό βρίσκει μέγα μέρος των Ευρωβουλευτών το πρόγραμμα για την διανομή τροφίμων στους πλέον απόρους της Ένωσης, ιδίως σε μια περίοδο κρίσεως ειδινών όπως αυτή που βιώνουμε σήμερα. Οι άνεργοι, οι κοινωνικά αποκλεισμένοι, οι άποροι αναμένουν αλληλεγγύη από την Ευρώπη με πρακτικούς και ξεκάθαρους τρόπους. Το βασικό μέσο για την παροχή υποστήριξης στα πιο ευάλωτα μέλη της κοινωνίας θα ήταν ένα ισχυρό Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει έναν εγγυημένο ελάχιστο προϋπολογισμό της τάξης του 25% της πολιτικής συνοχής και 20% της συνεισφοράς κάθε χώρας μέλους για τους κοινωνικούς αποκλεισμένους. Επίσης προτείνουμε να διατηρηθεί και να ενισχυθεί το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για να μπορεί να προσφέρει συγκεκριμένη αλληλεγγύη στους πρόσφατα ανέργους. Το πρόγραμμα της Κομισιόν για την υποστήριξη των πλέον απόρων στην Ευρώπη θα πρέπει να αποτελέσει μέρος της προσπάθειας αυτής. Η σκληρή πραγματικότητα είναι ότι πάντοτε θα υπάρχουν άνθρωποι στις κοινωνίες μας που θα έχουν ανάγκη από τέτοια προγράμματα. Και γι' αυτό στο κοινό δημοσιονομικό πλαίσιο 6 προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την βοήθεια σε τρόφιμα στον τίτλο 1 και μέσα στα πλαίσια της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Και αυτό είναι και ο καλύτερος τρόπος για να ξεπεραστούν τα νομικά εμπόδια που αντιμετώπισε το προηγούμενο πρόγραμμα. Όπως γνωρίζετε, οι συζητήσεις μεταξύ των χωρών μελών για την νομική βάση του τρέχοντος προγράμματος αντιμετώπισαν δυσκολίες. Η Κομισιόν χρειάστηκε να το σημειώσει βέβαια αυτό, αλλά δεν παρετείται του δικαιώματος πρωτοβουλίας της. Συμπεραίνοντας, κατά τη γνώμη μας, ο κοινοτικός προπολογισμό μπορεί να στηρίξει την διανομή τροφίμων και στο μέλλον στα πλαίσια μιας ευρύτερης προσπάθειας καταπολέμησης της φτώχειας. Και θα αναζητήσουμε διάφορους τρόπους για τη διαμόρφωση των μελλοντικών προγραμμάτων μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με συμμετοχή των διαφόρων ταμείων της συνοχής. Χρειαζόμαστε κάποιο χρόνο ακόμη για να καταστρώσουμε ένα πρόγραμμα που να είναι και αποτελεσματικό και ρεαλιστικό. Ευχαριστώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την συμβολή του και στην προσπάθεια και για το ότι έθεσε το θέμα προς συζήτηση. Τώρα θα λάβουν το λόγο οι πολιτικές ομάδες και πρώτος από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ο κύριος Σικίερσκι. Δύο λεπτά κύριε. Έχουμε, ε, αποφασίσαμε πέρσι σε δεύτερη ανάγνωση το πρόγραμμα διανομής τροφίμων στους αφόρους να συνεχιστεί για το 2012 και 2013. Στο τέλος δηλαδή της δημοσιονομικής προοπτικής. Στην συζήτηση για το μέλλον του προγράμματος, το πρόγραμμα βρήκε σημαντική υποστήριξη για την συνέχιση διανομής τροφίμων στους απόρους Τον δε Ιούλιο εγκρίθηκε ψήφισμα το οποίο διαλάμβανε τα εξή Ζητούσε να βρεθεί λύση για να μπορέσει να συνεχιστεί το πρόγραμμα υπέρ των πλέον απόρων στην Ευρώπη. Και για την επόμενη περίοδο 2014-2020 θα πρέπει να μπορεί να βασίζεται σε νομική βάση ώστε να μπορέσει να συνεχιστεί το πρόγραμμα και να μπορέσει να συνεχιστεί σε ικανοποιητικό βαθμό η διανομή τροφίμων έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι που εξαρτώνται από αυτή τη διανομή τροφίμων θα λαμβάνουν αρκετά. Και πριν από την ψηφοφορία μας στις 15 Φεβρουαρίου ο Επίτροπος Άντορ απάντησε σε ερωτήσεις της κυρίας Μπερές της Επιτροπής Απασχολήσεως σχετικά με το μέλλον του προγράμματος στην επόμενη δημοσιονομική περίοδο. Ο Επίτροπος Άντορ απάντησε λοιπόν λέγοντας ότι στο επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο θα χρηματοδοτηθεί το πρόγραμμα από άλλο τμήμα του προϋπολογισμού. Και διατύπωσε την άποψη ότι ο στόχος αυτός εντάσσεται και στους στόχους της Ευρώπης 2020 για την καταπολέμηση της φτώχειας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει χρήση του δικαιώματός της για να θέσει το θέμα στι διαπραγματεύσει για τον προπολογισμό. Οι δηλώσει του Επιτρόπου τη 21 η Δεκεμβρίου επίσης είναι σημαντικές για το προκείμενο θέμα. Οι αντίθετοι με το πρόγραμμα τελικά δήλωσαν διατεθειμένοι να αναζητήσουν συμβιβασμό στο Συμβούλιο και εμείς θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να λάβει υπόψη της τις χώρες οι οποίες δεν θέλουν να συνεχίσει το πρόγραμμα. Οι εργασίες συνεχίζονται. Πρέπει να γίνει και μια δημοσιονομική πρόταση συγκεκριμένη για το πρόγραμμα αυτό. Ευχαριστώ. Θα σας παρακαλούσα να τηρείτε το χρόνο γόρευσή σας. Και τώρα Εξ του των Σοσιαλιστών, το λόγο έχει η κυρία Μπερές, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με τον συνάδελφο Ντεκάστρο από την Επιτροπή Γεωργίας και ως πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων θελήσαμε και πάλι να φέρουμε το ζήτημα αυτό στην Ολομέλεια δεδομένων και των πρώτων δηλώσεων που έγιναν στις 15 Φεβρουαρίου εξ ονόματος του συνόλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλαδή επρόκειτο και προτίθεται να ε, ασκήσει το δικαίωμα πρωτοβουλίας για να κάνει μια πρόταση που θα επιτρέπει να χρηματοδοτήσει και το πρόγραμμα αυτό στο πλαίσιο των επομένων δημοσιονομικών προοπτικών. Στην πρωτοβουλία σε αυτή θα έχετε την πλήρη στήριξη του Κοινοβουλίου και το γνωρίζετε. Σας ζητούμε όμως να κάνετε ένα βήμα παραπάνω, γιατί αυτό το πρόγραμμα δεν μπορεί να είναι όμοιρο των διακυβερνητικών ε, διαπραγματεύσεων για την κοινή γεωργική πολιτική, ούτε να ακολουθεί κατά γράμμα ε, τις ε, αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων χωρίς να κυριαρχήσουν και πάλι νομοθετικές πρωτοβουλίες. Ζητούμε λοιπόν το πρόγραμμα αυτό να είναι γνήσιο πρόγραμμα αλληλεγγύης, δηλαδή να μην έρθει να να αντλήσει πόρους από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, γιατί αυτό που διοργανώνουμε έτσι είναι η αλληλεγγύη των φτωχών με τους φτωχούς και δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Σας ζητούμε κύριε Επίτροπε να προσέξετε το εξής. Εδώ στο Κοινοβούλιο πολλοί υποστηρίζουν όχι τη μακροοικονομική αιρεσιμότητα, εκεί δεν σας υποστηρίξουμε, αλλά τη θεματική αιρεσιμότητα και συγκέντρωση. Στη στρατηγική όμως για την Ένωση το 2020 έχετε ως στόχο την καταπολέμηση της ένδυας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Και θα πρέπει ε, οπωσδήποτε ε, ε, αυτό να απορρέει από κοινοτική χρηματοδότηση, από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Και θέλουμε και πιστεύουμε να πείσετε τα κράτη-μέλη. Μην τα μετράτε ε, τα κράτη ποια είναι υπέρ, ποια είναι κατά. Προσπαθήστε να τα πείσετε για να κινηθούν οι καταστάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα εξ των φιλελευθέρων κυρία Χάρκιν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχά να σα πω ότι καλωσορίζω τι προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα μεταβατικά μέτρα για να ε, βεβαιωθούμε ότι θα συνεχιστεί η χορήγηση τροφίμων στα πλέον άπορα άτομα στην Ένωση. Σήμερα 13 εκατομμύρια άποροι ε, σε 19 κράτη-μέλη που πλήττονται από τη φτώχεια δέχονται αυτή την υποστήριξη. Αυτό δείχνει πόσο μακριά πρέπει να φτάσουμε στην ανακούφιση τη φτώχεια. Είναι τεράστιε οι προκλήσεις που έχουμε ακόμα να αντιμετωπίσουμε. Και ενώ η παροχή τροφίμων από μόνη τη βέβαια δεν φτάνει για να ανακουφίσει τη φτώχεια, μπορεί να είναι ένα κομμάτι του πάζελ και για εκείνου που έχουν πρόσβαση σε αυτή τη βοήθεια είναι πραγματικά ουσιαστική. Συμφωνώ με τον Επίτροπο Ρεν ότι εκείνοι που ε, πρόκειται να πληγούν ή πλήττονται από τη φτώχεια, αναμένουν κάποια στοιχειώδη ελεγγύη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άκουσα τα σχόλια για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση. Δυστυχώ πολλά κράτη-μέλη δεν συμφωνούν μαζί σα. Οκτώ, νομίζω, δήλωσαν ότι θα πρέπει να καταργηθεί το Ταμείο αυτό. Ενώ υπάρχει υποστήριξη λοιπόν τη Κομισιόν και του Κοινοβουλίου για τη συνέχιση του Ταμείου αυτού, δυστυχώ δεν είναι αντίστοιχη η υποστήριξη από το Συμβούλιο. Επίσης φαίνεται ότι το πρόγραμμα που συζητούμε σήμερα αντιμετωπίζει δυσκολίες στο Συμβούλιο και θέτει το ευρύτερο ε, ζήτημα του μέλλοντος της κοινωνικής πολιτικής. Συμφωνούμε όλοι ότι μία από τις πέντε προτεραιότητες της στρατηγικής για το 2020 είναι η μείωση της φτώχειας. Ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποστηρίξει το Κοινοβούλιο. Και όπως γνωρίζετε είμαστε στο πλευρό σας κύριε Επίτροπη για το πρόγραμμα αυτό. Σας ευχαριστούμε. Επόμενη ομιλήτρια, εξ ονόματος των Πρασίνων, η κυρία Κορνέλησεν. Ένα μισή λεπτό έχετε στη διάθεσή σας. Πρόεδρε, καταφέραμε να διασφαλίσουμε ότι τα προγράμματα, τα επιστημιστικά δεν σταματήσαν για τα 80 εκατομμύρια απόρων που εξαρτώνται από αυτά και συνεχίζονται για το επόμενο χρόνο. Τώρα θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει σαφήνεια για το μέλλον. Το χειρότερο σενάριο είναι να συνεχίσουμε να δίνουμε την ιδέα στις τράπεζες τροφίμων. Το πρόγραμμα θα συνεχίσει μετά το 2014 και τελικά να ανακαλύψουν στη τελική φάση ότι δεν πρόκειται να συνεχιστούν. Αν δεν υπάρχει σαφήνεια τώρα, οι τράπεζε τροφίμων δεν θα πάρουν τα απαραίτητα μέτρα για να ε, σταματήσουν την εξάρτησή του από την ε, αρρωγή την ευρωπαϊκή. Είμαι βέβαιη ότι θα υπάρξει πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο για να συνεχιστεί αυτή η βοήθεια κατά κάποιο τρόπο. Αλλά επίση είμαι σίγουρη ότι θα υπάρχει πλειοψηφία στο Συμβούλιο που θα μπλοκάρει αυτή την απόφαση. Θα μπορούσε ο να Μα επιβεβαιώσει ότι η συμφωνία στο Συμβούλιο σημαίνει ότι θα μπορέσει να συνεχίσει το πρόγραμμα για δύο χρόνια, αλλά υπό τον όρο ότι θα σταματήσει μετά από αυτά τα δύο έτη και θα μπορούσε να μας πει ο Επίτροπος κατά πόσον υπάρχει ένας τρόπος να ξεπεράσουμε αυτό το μπλοκάρισμα, αυτό το φραγμό ή κατά πόσον ε, θα υπάρχει απλά η ελπίδα για κάτι καλύτερο, γιατί το να ελπίζουμε για το καλύτερο είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να προσφέρουμε από πλευρά βεβαιότητα στις ε, τράπεζες ε, τροφίμων και νομίζω ότι τελικά θα είναι ει βάρο τους αν δεν διευκρινίσουμε ότι θα σταματήσει το πρόγραμμα το 2014 προκειμένου να έχουν τουλάχιστον κάποιο χρόνο να προσαρμοστούν στο μέλλον. Σα ευχαριστώ και η επόμενη ομιλήτρια είναι η κυρία Τσίμερ για την Ενωμένη Ευρωπαϊκή Αριστερά. Δύο λεπτά έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, κύριε Επίτροπε, αν σωστά κατάλαβα, η δήλωση που κάνετε σήμερα ότι η νέη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αγωνίζεται για τη συνέχιση του προγράμματος αυτού, για τους απόρους της Ένωσης και ότι θα κάνει τα πάντα προκειμένου να υπάρξουν συγκεκριμένες προτάσεις εν ευθέτω χρόνο για το πού θα συνεχίσει το πρόγραμμα και ποια θα είναι η χρηματοδότηση. Νομίζω ότι αυτό είναι απαραίτητο πραγματικά. Και νομίζω ότι από κοινού είμαστε υπεύθυνοι προκειμένου να φροντίσουμε ότι το πρόγραμμα αυτοτροφίμων θα γίνει πραγματικότητα. Όχι. Γιατί αποτελεί ένα μήνυμα προς τον κόσμο ότι έχουμε ε, και καταλαβαίνουμε ε, την κατάστασή τους, καταλαβαίνουμε τις βασικές τους ανάγκες που δυστυχώς ε, μάλλον τις ανάγκες εκείνων που δεν μπορούν να συμμετάσχουν στην ανάπτυξη, που είναι τα μεγαλύτερα θύματα σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της ε, κρίσης ε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχω υπόψη μου την Ελλάδα, την Ισπανία, όλες αυτές τις άλλες χώρες όπου αυτά που πράττουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι εις βάρος των πλέον απόρων. Δίνουμε ένα μήνυμα, αλλά τίποτα παραπάνω. Νομίζω λοιπόν ότι είναι κατεπηγόντως απαραίτητο όχι μόνο να το δείξουμε αυτό στα 18 εκατομμύρια άτομα που εξαρτώνται από τα τρόφιμα που τους διατίθενται αυτά. Αλλά ότι το θέμα είναι ότι θέλουμε να συνεχίσουμε να καταπολεμούμε την ενδιά και ότι αυτό είναι στην κορυφή της των προτεραιοτήτων μας. Αυτό το μήνυμα δεν έχει ε, δοθεί ακόμη και αυτό είναι το πλέον καθοριστικό θεωρώ αν θέλουμε να σημειώσουμε πρόοδο, αν θέλουμε να μας εμπιστεύονται οι πολίτες, να εμπιστεύονται την Ευρωπαϊκή μας Ένωση, νομίζω ότι χρειάζεται μια κοινωνική και αλληλέγγυα Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν έχετε την υποστήριξή μας, αλλά οι συνάδελφοι εκλήθησαν να κάνουν κάτι προκειμένου ε, οι περιοχές, οι χώρε εκείνε οι οποίε μπλοκάρουν την κατάσταση να σταματήσουν να την μπλοκάρουν. Νομίζω ότι και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο. Ο κύριος Συμπράσα, επόμενος ομιλητής για το EFD. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η επιστημική κρίση και το αυξανόμενο κόστος διαβίωσης αναγκάζουν όλο και πιο πολύ κόσμο να εξαρτάται από την αρρωγή αυτή. Για το 2012 ε, το πρόγραμμα αυτό ε, θα ανέλθει στα 113 εκατομμύρια και αυτό αποτελεί μεγάλη μείωση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, περίπου 43 εκατομμύρια ε, κόσμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να φροντίσει για τις καθημερινές επιστηστικές του ανάγκες. Και οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις τονίζουν πόσο σημαντικό είναι το πρόγραμμα επιστημιστικής αρρωγής. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να βρεθεί μία λύση χωρίς να περιοριστούν ε, τα ποσά χρηματοδότησης. Και επίσης το αυξανόμενο κόστος θέρμανσης ε, υπογραμμίζει ακόμα πιο πολύ την έντονη ανάγκη που έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Και στη Λουθιανία αυτό πραγματικά επηρεάζει πάρα πολύ κόσμο. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενη ομιλήτρια, η κυρία Μορβάη, για τους μη κυγραμμένους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Το σύστημα παροχής ε, τροφίμων στους απόρους δεν βοηθάει μόνο εκείνους τους απόρους που είναι οι τελικοί αποδέκτες, αλλά και τις εταιρείε που με το σύστημα των δημοσίων προμηθειών αποκομίζουν μεγάλα κέρδη. Και δεν είναι άσχετο ούτε αδιάφορο το ποιες, ποιες εταιρείε είναι αυτές. Θα παρακαλέσω τους βουλευτές να κοιτάξουν στις χώρες τους ποιες εταιρείε παίρνουν αυτά τα χρήματα. Τα αποτελέσματα είναι ε, πραγματικά εντυπωσιακά. Στην Ουγγαρία έχουν δοθεί πάρα πολύ μεγάλα ποσά ε, για αγορά τέτοιων τροφίμων και πηγαίνουν στις μεγάλες επιχειρήσεις και όχι στις μικρομεσαίες γύρω στα 4 δις. 660 εκατομμύρια έχει πάρει μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στη Ουγγαρία. Και αυτές οι επιχειρήσεις έχουν ε, καταδικαστεί ε, για ε, δημιουργία καρτέλ. Πάντα υποστηρίζουμε τις μικρομεσαίες στα λόγια και αντί γι' αυτό τα δημόσια κονδύλια πηγαίνουν στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στα κράτη-μέλη. Καλό θα ήταν λοιπόν να υποφελούνται και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να έχουν την αίσθηση ότι δεν είναι πάντα χαμένοι επειδή δεν βρίσκονται κοντά στην εκάστοτε κυβέρνηση. Τουλάχιστον στην Ουγγαρία αυτή την αίσθηση έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν στηρίζονται. Στηρίζονται μόνο αυτές που είναι φίλοι του καθεστώτος. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σιλβέστρης τώρα. Ακολουθούν οι μεμονωμένοι μελητέ. Παρακαλώ. 18 εκατομμύρια εξαρτώνται στην Ευρώπη από το πρόγραμμα αυτό. Και 43 ε, εκατομμύρια πολιτών κινδυνεύουν να πέσουν στη φτώχεια. Ευχαριστώ τον συνάδελφο Σικέρσκι και τους υπολείπου που ε, ασχολήθηκαν με αυτό το θέμα στι αρμόδιες επιτροπές. Αλλά θα πούμε αμέσω ότι απορρίπτουμε την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής ω προ το προσωρινό του προγράμματος. Δεν είναι ε, σωστό αυτή η ιδέα ότι η έγκριση και η συμφωνία θα πρέπει να έρθει ε, ε, από το Συμβουλίο Γεωργίας όπως συμφωνήθηκε στις 14-15 Δεκεμβρίου να σταματήσει το πρόγραμμα. Αυτή η ιδέα είναι κάτι που απορρίπτουμε ήδη. Αν υπερψηφίσουμε σήμερα θα κάνουμε μια προσπάθεια από αύριο για να επαναδραστηριοποιηθεί, να κινητοποιηθεί το πρόγραμμα. 2,5 δισεκατομμύρια ε, υπάρχουν στο αποθεματικό των επομένων δημοσιονομικών ε, προοπτικών για την περίοδο 14-19 στις κοινωνικές υποθέσεις. Μπορεί λοιπόν με την ισχύα της Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει συνέχεια σε αυτό το πρόγραμμα και να διατρανώσει και πάλι ε, την πρόθεσή της να συνεχιστεί το θέμα. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη από βοήθεια στην Ευρώπη που πλήττεται και υποφιλείται αυτό το πρόγραμμα. Δεν μπορεί ε, με φόρους και περικοπές ε, η Ευρώπη να αντιμετωπίσει την κρίση χωρίς να βοηθάει τους απόρους. Αυτή είναι μια ε, κοντόφθαλμη πολιτική. Από αύριο λοιπόν, αφού θα έχουμε εγκρίνει το πρόγραμμα, θα αγωνιστούμε για να συνεχιστεί και μετά το 2014. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητή ο κύριο Δεκάστρο, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αξιότιμοι συνάδελφοι, θα ήθελα καταρχά να θυμίσω ε, με έντονη ικανοποίηση το πολύ σημαντικό αποτέλεσμα που καταφέραμε να επιτύχουμε με την ε, παράταση για το 2013 του παρόντος προγράμματος. Ήταν μακρά και δύσκολη η πορεία ε, όπου στρατεύτηκε όλο το Κοινοβούλιο. Τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή μάλλον η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και η Επιτροπή Γεωργίας από κοινού ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δεσμευτεί ρητά ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη συνέχιση του προγράμματος μετά το 2013. Στι 6 Δεκεμβρίου έκανε μια ανακοίνωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπου ελάμβανε υπόψη τι δυσκολίε των νέων κρατών μελών. Δεν μπορεί όμω να προεξοφλήσει αυτό το δικαίωμα νομοθετική πρωτοβουλίας Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπω προβλέπεται στη συνθήκη. Η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη της την έντονη βόληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ε, την ευρύτατη πλειοψηφία των κρατών μελών τη Ένωση που επιθυμούν τη συνέχιση του παρόντος προγράμματο και εμεί διαπιστώνουμε και σημειώνουμε με ικανοποίηση τι σημερινέ δηλώσει Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θυμίζουμε ακόμα ότι το εργαλείο που δίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη δυνατότητα ε, να δίνουν 440 ε, εκατομμύρια ε, ποσότητες τροφίμων και σε οικογένειες και σε παιδιά στην Ένωση είναι μια πολιτική πρωτοβουλία. Το ξέρουμε κύριε Επίτροπε ότι υπάρχουν παγκόσμιες προκλήσεις. Ε, αλλά αυτές οι παγκόσμιες προκλήσεις επιτείνουν τις δυσκολίες των πιο φτωχών και των απόρων. Ελπίζουμε από το 2014 και μετά να συνεχιστεί το πρόγραμμα αυτό. ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βουλευτά. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Λάιον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Το πρόγραμμα αυτό <clears throat> είχε δημιουργηθεί σε μια εποχή που υπήρχαν διατροφικά πλεονάσματα στην Ευρώπη. Τώρα αυτό δεν ισχύει πλέον. Τώρα η Κομισιόν αγοράζει από την αγορά τρόφιμα για να τα δώσει στους πλέον απόρους. Και το δικαστήριο εξέθεσε σε απόφαση αντίθετη, γι' αυτό πρέπει να βρούμε άλλους τρόπους. Το κόμμα μου θεωρεί ότι Πρέπει να βρεθούν τρόποι για να βοηθηθούν οι πλέον άποροι στην Ευρώπη και αυτό, σε αυτό συμφωνούν όρισμένε χώρε μέλη στο Συμβούλιο. Ωστόσο, η ΚΑΠ δεν αποτελεί πλέον το κατάλληλο εργαλείο για να στηριχθεί το πρόγραμμα στο μέλλον. Γι' αυτό και στηρίζω την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην επόμενη δημοσιονομική περίοδο <clears throat> να ληφθεί το Κοινωνικό Ταμείο ως βάση και η απόφαση του δικαστηρίου επιτρέπει μια εθνική ευελιξία στο θέμα αυτό. Και έτσι θα μπορέσουμε να στηρίξουμε τους πλέον άπορους πολίτες στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ντελή. C'est bon là? Εντάξει τώρα. Κύριε Επίτροπε, η πρόταση Γενικού Κανονισμού για τα Διαρθρωτικά Ταμεία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής προβλέπει 5 δισεκατομμύρια ευρώ για τη μελλοντική διατροφική βοήθεια για την περίοδο 2014-2020 και παρά την πεισματωμένη αντίσταση, αντίσταση ορισμένων χωρών στο Συμβούλιο. Η πλειοψηφία των χωρών δέχεται αυτό που ζητεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και βέβαια η πλειοψηφία των πολιτών μας, οι οποίοι όλοι και περισσότερο στρέφονται στις τράπεζες τροφίμων σε ολόκληρη την Ευρώπη λόγω της επιδείνωσης της κοινωνική κρίσης. Είναι θαραλέο, αλλά δεν είναι αρκετό. 500 εκατομμύρια ευρώ, το πολύ. Ενώ έχουμε 2,5 δισεκατομμύρια στον προϋπολογισμό για τα πράγματα αυτά. Μείωσε η Κομισιόν κατά ένα δισεκατομμύριο, παρόλο που οι ανάγκες είναι όλο και περισσότερε. Δεν γνωρίζουμε και τίποτε για τις προθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καθιέρωση του μελλοντικού προγράμματος. Και θα είναι μέσα στα πλαίσια του μηχανισμού στήριξης θα μπορούν με τη βάση αυτή να αγοράζουν από την αγορά γεωργικών προϊόντων τρόφιμα για να τα διανύμουν στους ε, απλέον απόρους ενώ υπάρχει και αντίθετη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου οι τράπεζες τροφίμων κινδυνεύουν να βρεθούν στην ίδια θέση από αυτήν που μόλις τώρα κατάφεραν να ξεφύγουν. Τι προεκτίθεστε να κάνετε. Εγώ θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει ένας ικανοποιητικός προϋπολογισμός για το πρόγραμμα αυτό, να διασφαλιστεί ότι ο κάθε ένας και κυρίως οι πλέον άποροι να έχουν εξασφαλισμένη μια υγιεινή διατροφή και να υπάρχει και ένα δίχτυ ασφάλειας με μια πραγματική οδηγία Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ομαργή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Λυπούμε, διότι δεν μπορέσατε να μας ανακοινώσετε τίποτα το συγκεκριμένο. Είπατε ότι θα βασιστείτε στο κοινωνικό ταμείο, αλλά χωρίς να το αυξήσετε. Εάν βάλετε 2,5 δισεκατομμύρια σε ένα πολιετές πρόγραμμα αφιερωμένο στον τομέα αυτό, είτε το θέλουμε είτε όχι, αυτό σημαίνει ότι θα μειωθεί κατά 100 εκατομμύρια ευρώ το ποσό που διατίθεται κάθε χρόνο σε αυτή την ε, επιστημιστική βοήθεια. Δεν μπορούμε να δεχθούμε εμείς την κατάσταση αυτή. Γι' αυτό προτείνω Κοινοβούλιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβουν κοινή πρωτοβουλία, μια κοινή δηλαδή συνεδρίαση με τις οργανώσεις αλληλεγγύης στην Ευρώπη, για να αξιολογηθούν ακριβώς οι ανάγκες τους και σε νούμερα δηλαδή και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στη συζήτηση με όλα αυτά τα νομικά εργαλεία. Ευχαριστώ η κυρία Μωρόν Σατιέ. μισή λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, παρακολούθησα την παρέμβασή σας. Προτείνετε το πρόγραμμα βοήθειας να βασιστεί στο κοινωνικό Ταμείο. Υπενθυμίζω κύριε Επιτροπέ ότι το Κοινωνικό Ταμείο στο μεγαλύτερο μέρος του κατευθύνεται στην επαγγελματική ένταξη η οποία όμως επαγγελματική ένταξη είναι το απολύτως απαραίτητο εργαλείο για την κοινωνική ένταξη. Δεν, υπάρχει, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει κοινωνική ένταξη χωρίς επαγγελματική. Θα χρειαστεί λοιπόν να συνεχίσουμε τις, την επαγρύπνησή μας για την επαγγελματική ένταξη. Για τα προγράμματα τώρα παροχής τροφίμων στους πλέον απόρους, εμείς θεωρούμε ότι τα ποσά που έχουν μέχρι κατανεμηθεί τώρα, δηλαδή 500 εκατομμύρια ευρώ ανά έτος, να παραμείνουν τουλάχιστον μέχρι το 2020. Ναι, θα χρειαστεί να πείσετε τις τακτικές χώρες, αυτές που σήμερα εκφράζουν επιφυλάξεις αλλά δεν μπορούμε να βάλουμε απλώς ρήτρα αιρεσιμότητας στα κοινωνικά προγράμματα. Έχουμε ανάγκη των προγραμμάτων αυτών. Εμείς κινητοποιούμεθα για να το υπερασπιστούμε και εσείς έχετε την ευθύνη να εξασφαλίσετε τη διάρκεια του. Ευχαριστώ πολύ, ο Πρόεδρος. Ο κύριος Ντάντα για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, έχουμε επαναλάβει έχουμε πει κατ' επανάληψη εδώ ότι αν δεν δώσουμε περισσότερα μηνύματα αλληλεγγύης στους πολίτες ότι συμπαρατάσσεται μαζί τους δηλαδή η ε, Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί τους αυτοί θα μακριθούν ακόμη περισσότερο όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει μια μειοψηφία που μπλοκάρει κάθε σχετική πρωτοβουλία στο Συμβούλιο και δεν είναι το μοναδικό παράδειγμα και το Ταμείο προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση υπέστη τα ίδια. Ωστόσο, έχετε αναλάβει μια πρωτοβουλία για να διασώσετε το σημαντικό αυτό πρόγραμμα και να γίνει ένα πρόγραμμα διαρκού αλληλεγγύη. Αυτά είναι μηνύματα που αναμένουν οι πολίτε. Μην χαθεί αυτή η ευκαιρία, μην διστάσετε. Οφείλουμε να πείσουμε το Συμβούλιο και εν πάση περιπτώσει τουλάχιστον μέχρι να έρθουν στο Συμβούλιο η γερμανική και η γαλλική σοσιαλιστική κυβέρνηση. Ο κύριος Χόισλινγκ τώρα για ένα λεπτό. Νομίζω ότι διακομματικά συμφωνούμε και θα μπορέσουμε να πείσουμε τις χώρες οι οποίες αντιτίθενται μέχρι τώρα στην συνέχιση του προγράμματος. Καθήκον μας είναι να φανούμε αλληλέγγυοι με τα 18 εκατομμύρια ανθρώπων που έχουν ανάγκη από το πρόγραμμα. Αλλά βέβαια πρέπει να βασιστεί σε νέα βάση. Αυτό είναι σαφέ, διότι τα πλεονάσματα, σωστά τα είπε προηγουμένω ένα συναδελφό μου, δεν υπάρχουν πλέον τα πλεονάσματα τη κοινή αγροτική πολιτική. Γι' αυτό πρέπει να βρούμε άλλο τρόπο. Λαμβάνοντα υπόψη βέβαια και τι αποφάσει του δικαστηρίου. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να ενισχύσουμε τι περιφερειακέ πρωτοβουλίε και αυτές διανομής τροφίμων και αυτές που υποδέχονται τρόφιμα από διάφορους δωρητές. Πρέπει όμως να υπάρχει μια εξασφάλιση της διάρκειας. Δεν μπορούμε να μιλούμε κάθε φορά ξανά για μόνο για μια διετία. Οι άνθρωποι που εξαρτώνται από τις διανομές τροφίμων έχουν ανάγκη από την εξασφάλιση αυτή και μάλιστα μακροπρόθεσμα. Ευχαριστώ. Τότε κυρία Τσούμπρη για ένα λεπτό έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Η σημερινή κοινωνική κατάσταση είναι πραγματικά παράδεκτη 43,3% πάνω από 15 εκατομμύρια Ευρωπαίοι είναι στο όριο της φτώχειας και ακόμα και οι εργαζόμενοι απειλούνται από τη φτώχεια. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, ε, το, κίνδυνος ένδυας θα πρέπει να θεωρηθεί σε σχέση και με τις κακοπληρωμένες και επισφαλείς θέσεις ε, εργασίας και σε ό,τι αφορά τον προπολογισμό που αποφασίστηκε στο Κοινοβούλιο, ε, θα επιδεινώνει περαιτέρω την κατάσταση. Δεν είναι πραγματικά αποδεκτό αυτό σε τέτοιους δύσκολους καιρού ε, να σταματήσει το πρόγραμμα αυτό για τους άπορους και για τους εργαζόμενους αυτούς. Ένα πρόγραμμα το οποίο έχει να κάνει με την επιστημιστική ασφάλεια. Θα ήταν ασφαλώς καλύτερο να είχαμε μεγαλύτερο ποσό από τα 500 εκατομμύρια που προτείνονται, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συνεχιστεί το πρόγραμμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ένα μισή λεπτό τώρα η κυρία Χεράντ Γκαρσία. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, χάρη στη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τράπεζες τροφίμων κάνουν κοινωνικό έργο αξιέπαινο που έχει αναγνωριστεί και θα πρέπει να μπορεί να συνεχιστεί στο μέλλον με την αναφυσβήτητη υποστήριξη του Κοινοβουλίου. Μια από τις βασικές και θεμελιώδεις αρχές της Ένωσης είναι η ε, κοινωνική συνοχή, η εδαφική συνοχή και αλληλεγγύη. Και αυτό είναι αμέτροπο στην κατεύθυνση αυτή η κρίση μαστίζει τους Ευρωπαίους πολίτες. 80 εκατομμύρια βρίσκονται κάτω από το κατόφλι της φτώχειας και 43 εκατομμύρια σκέφτονται πολύ αν θα φάνε πρωτεΐνες πάνω από δύο φορές την εβδομάδα ή μάλιστα δύο φορές την εβδομάδα η κοινή γεωργική πολιτική θα πρέπει να συμμετέχει και στην προσπάθεια αυτή. Ω βουλευτέ θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προωθήσουμε τι πρωτοβουλίε έτσι ώστε να συνεχιστεί το πρόγραμμα αυτό από το 2014 και μετά και καθ' όλη την επόμενη προγραμματική περίοδο των δημοσιονομικών προοπτικών από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να επιβάλλουμε συμφωνία στο Συμβούλιο ε, Υπουργών και θα πρέπει να αφήσουμε στην άκρη τους ε, εγωισμούς και να σκεφτούμε τους Ευρωπαίους πολίτες. Σας ευχαριστώ πολύ. Επόμενη ομιλήτρια, 1,5 λεπτό κύριε Σάρμπουλ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Η συμφωνία η οποία συνάφθηκε μετά από τις διαθεσμικές διαπραγματεύσεις ε, προβλέπει ότι το πρόγραμμα ε, τροφίμων θα συνεχιστεί με την ίδια χρηματοδότηση μέχρι το 2013. Δυστυχώς, κάποια κρατημέλη τάχθηκαν υπέρ της κατάργησης του προγράμματος ολοσχερός μετά το 2013. Πάνω από 18 εκατομμύρια πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνουν τρόφιμα μέσω του προγράμματος αυτού. Και ας μην ξεχνάμε ότι πάνω από 18 εκατομμύρια Ευρωπαίοι ζουν κάτω από το όρο της ένδυας. Θα ήθελα να υπογραμμίσω το εξή, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η πείνα και η ένδυα υπάρχουν και στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορούμε να τα γνωρούμε αυτά. Και όλα αυτά έχουν επιτυνευθεί με την οικονομική κρίση η, τα αριθμητικά στοιχεία που ανέφερα ε, καταδεικνύουν πόσο σημαντικό θα είναι το πρόγραμμα αυτό και στο μέλλον. Θα είναι πραγματικά απάνθρωπο να σταματήσει ένα τέτοιο πρόγραμμα σε μία περίοδο η οποία μόνο χειρότερη μπορεί να γίνει. Δεν θα εξαφανιστεί η φτώχεια το 2013 και με εξή. Θα πρέπει να συνεχιστεί λοιπόν το πρόγραμμα αυτό και θα πρέπει να παραμείνει ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο θα χαίρει τη ίδια χρηματοδότηση όπω και τώρα. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δει πού μπορεί να εντάξει το πρόγραμμα αυτό σε ό,τι αφορά το επόμενο πολιτές ε, ε, χρηματοοικονομικό πλαίσιο και προτείνω να εισαχθεί η χρηματοδότηση. Οι συζητήσεις για το επόμενο πολιετές ε, χρηματοοικονομικό πλαίσιο συνεχίζονται, αλλά το θέμα του προγράμματος αυτού δεν έχει ακόμα επιληθεί. Δεν θα πρέπει όμως να αγνοηθεί το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Τελευταία ομιλήτρια, η κυρία Πατράου Νέβες. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Θα ήθελα να συγχαρώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί έχει διασφαλίσει πλέον ένα ε, κομμάτι του προπολογισμού για τους πλέον άπορους σε καιρούς ε, χρηματοοικονομικής κρίσης. Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση δραστηριοποιείται σε τομείς εξωτερικής πολιτικής, δεν ε, είναι αποδεκτό να μην συνεχίσει το πρόγραμμα παροχής ε, τροφίμων ύψους 500 εκατομμυρίων. Αλλά είναι περιορισμένο το πρόγραμμα αυτό, γιατί μετά το 2013 δεν υπάρχει οποιοδήποτε διασφάλιση ότι θα συνεχιστεί το πρόγραμμα αυτό. Τα κράτη-μέλη, τα οποία δηλώνουν ότι οι τράπεζες ε, τροφίμων θα πρέπει να λειτουργούν σε εθνική βάση, θα πρέπει να αναλογιστούν κατά πόσον ο πολιτικός, οικονομικός και οικονομικός χώρος είναι κάτι που έχουμε κοινό και θα πρέπει να μας βρίσκει αλληλεγγύους. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα θα δώσω το λόγο σε πέντε βουλευτές στα πλαίσια της διαδικασίας Catch the Ο κ. Δεμέιρα. Δίας ευχαριστώ Πρόεδρε. Αναλαμβάνω την ανάγκη να καταλήξουμε σε γενική συμφωνία στραμμένη στο μέλλον για να εξασφαλιστεί η επιβίωση των πιο πόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ευάλωτοι, αποκλεισμένοι, φτωχοί άνθρωποι. Από στοιχεία που έχουμε 13 εκατομμύρια φτωχών και σε 19 κράτη-μέλη και 30 εκατομμύρια υποσυντίζονται, ενώ 43 εκατομμύρια βρίσκονται σε επιστημιστική φτώχεια. Αυτό μας επιβάλλει συνεργασία για να καταφέρουμε συνέχιση του και διατήρηση του προγράμματος μετά το 2013. Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τη συζήτηση για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, καθώς επίσης και τη συζήτηση που γίνεται για την μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί αυτή η βοήθεια και να σταματήσουν τα νομικά εμπόδια. Τα κράτη-μέλη διανύουν περίοδο δυσκολιών, αλλά ακριβώς για αυτό το λόγο τώρα θα πρέπει να κάνουμε μεγαλύτερες προσπάθειες για να προστατεύσουμε εκείνους που πλήττονται περισσότερο από την κρίση. Τα παιδιά, τους ασθενείς, ε, τους ανέργους, τους ηλικιωμένους και γενικά 80 εκατομμύρια σήμερα ζουν κάτω από το κατόφλι της φτώχειας. Το δικαίωμα πρωτοβουλίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ζωτική σημασία και θεμελιώδες. Στο Κοινοβούλιο, κύριε Πρόεδρε, δεν διαφωνούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Τελείωσα. Ευχαριστώ, κυρία Ιρεγκόιεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, Επίτροπε, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το κακό στη ρίζα του, στην αιτία του το πρόβλημα. Και αυτό είναι το σημερινό φιλελεύθερο οικονομικό μοντέλο που εφαρμόζουν πολλά κράτη-μέλη με στρατηγικές που βασίζονται σε δημοσιονομικές προσαρμογές χωρίς όμως ενεργέ πολιτικές που να δημιουργούν ανάπτυξη και θέσεις απασχόλησης και συνδέονται με μια ανισορροπία και του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα που πλήττουν ε, τους πολίτες οι οποίοι δεν φταίνουν για την κρίση και τους ρίχνουν στη φτώχεια, στην πείνα και στον κοινωνικό αποκλεισμό. Πάνω από 113 εκατομμύρια πολιτών κινδυνεύουν να πέσουν στη φτώχεια στον κοινωνικό αποκλεισμό. Η αλληλεγγύη και η συνοχή είναι βασικέ αρχέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και μα υποχρεώνουν να διορθώσουμε αυτέ τι πολιτικέ και να ρυθμίσουμε τι οικονομικέ σχέσει για να μην αυξηθεί ακόμα περισσότερο η ψαλίδα των διαφορών και να υπάρξει μια ισορροπία. Η Ευρώπη θα πρέπει να είναι στο πλευρό των πολιτών, των πολιτών που πλήττονται περισσότερο για να τους δώσει μια ελπίδα για μια κρίση, έξοδο από την κρίση. Συγγνώμη. Μόνο έτσι θα ανακτήσει τη χαμένη της αξιοπιστία η Ένωση και χρειάζεται οπωσδήποτε να συνεχιστεί το παρόν πρόγραμμα. Ευχαριστώ ο Πρόεδρος, ο κύριος Κέλλη. Ε, σας ευχαριστώ και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να συζητήσουμε το θέμα αυτό, ιδιαίτερα μιας και είμαστε διάσημοι σε όλο τον κόσμο, θέλετε, για την παροχή ε, βοήθειας και επιστημικής ε, βοήθειας ιδιαίτερως. Εκ παραλλήλου, ωστόσο, θα πρέπει να τονίσουμε ότι πολλοί από τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρήζουν βοήθειας γιατί πλήττονται από την ένδυα, από τον κοινωνικό αποκλεισμό. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε λοιπόν να τους βοηθήσουμε. Είναι δική μας ευθύνη να τους χορηγήσουμε τη βοήθεια αυτή. Όχι μόνο φέτος και του χρόνου, αλλά μέχρι το 2020 για να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει στο σχέδιο αυτό και ελπίζουμε να συνεχιστεί το πρόγραμμα αυτό και μετά το 2020 άλλωστε. Θα πρέπει να συνεχιστεί λοιπόν και μελλοντικά το πρόγραμμα αυτό. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Κουέρες, για ένα λεπτό. Yes. Ο κύριος Γκερέρο, ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Πίτροπε, το ηθικό ανάστημα μιας κοινωνίας δεν μετριέται ουσιαστικά από το ΑΕΠ, μετριέται από τον τρόπο που δίνει μόρφωση στα παιδιά της, τον τρόπο που ε, ε, εξασφαλίζει την υγεία όλο το μέλλον, κυρίως πώς προστατεύει τους ε, ανθρώπους και τους πολίτες που είναι σε λιγότερο ευνοημένη θέση. Μπορεί να φέρετε μικρό το πρόγραμμα, αλλά δεν είναι καθόλου έτσι, διότι από το πρόγραμμα αυτό εξαρτάται η ηθική διάγνωση που θα βγάλουμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μόνο οικονομικό εγχείρημα και σχέδιο, είναι ένα σχέδιο συνεργασίας και αλληλεγγύης αλληλεγγύης με εκείνου που χρειάζονται περισσότερο την αλληλεγγύη μας. Όταν 43 εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών μας έχουν ανάγκη, η απόφαση δεν μπορεί να εξαρτάται από το ποια θα είναι η νομική βάση που θα εφαρμόσουμε. Δεν μπορούμε να χάνουμε χρόνο συζητώντας το διαδικαστικό. Γι' αυτό λοιπόν υποστήριζω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να υπερασπιστεί το ηθικό ανάστημα του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και αν ε, ε, δεν πρόφερα σωστά το όνομά σας, ε, πολύ λυπάμαι και ζητώ συγγνώμη. Mm. Τελευταίος ομιλητής, ε, η τελευταία μάλλον ομιλήτρια. Η κυρία Ζολταν Σίσιλη, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να συνεχιστεί η διανομή τροφίμων μετά το 2008 μας βρίσκει σήμερα σε μια χειρότερη κατάσταση ακόμη από το 2008 γιατί είναι ακόμα πιο πολλοί άποροι, ακόμα πιο πολλοί αυτοί που πεινούν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να παραμείνει αλληλέγγυη θα πρέπει να εισαγάγουμε μέτρα τα οποία θα ενισχύσουν τους πλέον Να μην ξεχνάμε επίσης και αυτούς που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης. Θα πρέπει να τονίσω ότι στην χώρα μου, την Σλοβενία, σε κάποια τμήματα η κατάσταση είναι τόσο τραγική που ακόμα και οι οργανώσεις ε, οι φιλανθρωπικές σταμάτησαν τη διανομή τροφίμων γιατί δεν υπάρχουν πολύ απλά τρόφιμα για να διανέμουν. Τέτοια μέτρα λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πολύ ευπρόσδεκτα και θα πρέπει να συνεχιστεί η προσπάθεια αυτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ο, λέει ο πρόεδρο, και τώρα ο κ. έχει το λόγο για να ολοκληρώσει τη συζήτηση. Uh, Ευχαριστώ Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτέ. Θα ήθελα καταρχά να καλωσορίσω την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το πρόγραμμα αυτό. Όπως τα γνωρίζετε, 2,5 εκατομμύρια είχε προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο επόμενο πολίτες ε, χρηματοοικονομικό πλαίσιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το δικαίωμα πρωτοβουλία στον τομέα αυτό. Συμφωνώ ότι η αρρωγή στον τομέα των τροφίμων εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο καταπολέμησης της ένδυα στην κοινωνία και κατά πάσα πιθανότητα θα γίνει αποδεκτό μόνο εάν ε, συγκαταλέγεται μεταξύ άλλων συνεκτικών μέτρων για την καταπολέμηση της ένδυας κατά προτίμηση μέτρων που θα χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Σε ό,τι αφορά τα σχόλια διαφόρων βουλευτών, θα ήθελα να αναφέρω το εξής, ότι όντως θέλουμε να αγωνιστούμε προκειμένου να συνεχιστεί αυτή η επιστηστική αρρωγή και στο μέλλον, όπως προτείναμε άλλωστε, αλλά αντιλαμβανόμαστε επίσης ότι συντόμως θα πρέπει να ανακοινώσουμε είτε τη συμφωνία μας είτε την απόρριψη της συνέχισης του προγράμματος προκειμένου όλα αυτά τα προγράμματα και όλες οι τράπεζες τροφίμων να μπορέσουν να προσαρμοστούν. Όσοι ρωτούν τώρα γιατί θα πρέπει αυτό το πρόγραμμα να υπάρχει, σε αυτούς όλους απαντούμε το εξής, ότι σε μια εποχή που έχουν τεθεί κοινοί στόχοι, κοινά συμπεφωνημένοι στόχοι σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της ένδυας, η Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ απλά δεν μπορεί να αγνοήσει το γεγονός ότι παραπάνω από 43 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες δεν μπορούν να ε, έχουν ένα γεύμα με πρωτεΐνες κάθε δεύτερη μέρα, μέρα παραμέρα και ότι πολλά παιδιά δεν έχουν ε, το γάλα που χρειάζονται κάθε μέρα γιατί οι γονείς τους είναι φτωχοί. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη δεν πρέπει να θεωρηθεί μόνο ένα ιδανικό αλλά καθίσταται ηθική επιταγή. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ λέει και ο Πρόεδρος. Πέρα στη συζήτηση. következő και τώρα θα περάσουμε στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Είναι η